Την επόμενη έκθεση, έκθεση της κυρίας Γκρίσπεκ, τεκμήριο αθωότητας και δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινική διαδικασίας. Να δώσω καταρχάς το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Γκρίσπεκ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, παρόλο που η ώρα είναι προχωρημένη, χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να αναφέρω στο πλαίσιο της συζήτησης σήμερα αυτή την οδηγία για το τεκμήριο της αθωότητας, κάτι για το οποίο εργαζόμαστε εδώ και πολλούς μήνες και που τελικά ε, καταλήξαμε σε ένα αποτέλεσμα, ε, μια συμφωνία που ήταν δύσκολη αλλά που είναι μια καλή συμφωνία γιατί τελικά τρώνεται σε ένα κείμενο το οποίο είναι φιλόδοξο όσον αφορά τον σεβασμό των, ανθρωπίνων, των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Το, την 31η Μαΐου πέρσι μου δώσατε μια ξεκάθαρη αντολή. Η θάση του Κοινοβουλίου ήταν ε, ξεκάθαρη. Επιθυμούσε μια ε, μεγαλύτερη προστασία για τους ε, διοκόμενους ή τους κατηγορούμενους. Μια πρωτοβολία, μια, μια οδηγία η οποία να εναρμονίζει τι ε, εθνικέ νομοθεσίε, προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Είδου λοιπόν το περιεχόμενο αυτής της οδηγίας. Το δικαίωμα να μην κατηγορείται κανεί ε, δημόσια από τις ε, δημόσιες αρχές πριν από τη δίκη ε, σημαντικό ε, μετά τις ε, επιθέσεις στο Σαρλί Επτό όπου ένας φοιτητής κατηγορήθηκε ότι είχε συμμετάσχει στις επιθέσεις στα Άραβας ενώ ήταν απολύτως αθώος και ήταν στο πανεπιστήμιο. Και αυτή η εμπειρία ήταν εξαιρετικά τραυματική. Αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία προτίθεται να απαγορεύσει όλες τις δημόσιες δηλώσεις κρατικών αρχών που υπονοούν ότι κάποιο κατηγορούμενο είναι ένοχο πριν από την εξαγωγή τη δίκη. Και υπάρχει ένα ξεκάθαρο ορισμό στο κείμενο ε, των δημόσιων ε, δηλώσεων. Δεύτερον, πρόκειται για μια νίκη για το Κοινοβούλιο, γιατί η οδηγία περιλαμβάνει ένα νέο άρθρο για τον τρόπο με τον οποίο ε, θα πρέπει να παρουσιάζεται το ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να είναι μέσα σε ένα κλωβό και δεν μπορεί να είναι ε, τιμένος με τα ρούχα των ε, κατηγορουμένων ε, των φυλακισμένων ε, γιατί με τον τρόπο αυτό προδικάζεται το αποτέλεσμα της δίκης. Η οδηγία επίσης αναφέρεται στην αρχή του προωρέου, ε, βάσει τη κάθε αμφιβολία για την ενοχή ενό κατηγορουμένου θα πρέπει να είναι ει όφελός του. Και ε, εάν υπάρχουν αμφιβολίε, ο κατηγορούμενος θα πρέπει να, αθώ, να αθώνεται. Ε, ε πρόκειται για μια βασική αρχή του ποινικού δικαίου σε σχέση με το βάρος της απόδειξης. Ε, και μια βασική μάχη ήταν γύρω από την αντιστροφή του βάρους απόδειξης ε, όπου πραγματικά βάλαμε μια κόκκινη γραμμή και πετύχαμε το στοιχείο αυτό να μην ισχύει παρά μόνο σε πολύ περιορισμένες ε, ε, περιπτώσεις όπου υπάρχει ένα τεκμήριο ενοχής για τον ε, κατηγορούμενο. Πρόκειται λοιπόν για μια σημαντική εξέλιξη όπως και η προάσπιση του δικαιώματος σιωπή για τον κατηγορούμενο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα στοιχείο το οποίο οδηγεί στην υπόθεση της ενοχής του. Ο κατηγορούμενος έχει επίσης δικαίωμα να παρίσταται στη δίκη του και ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι τα αποδεκτικά στοιχεία ε, τα οποία ε, θα πρέπει ε, να συγκεντρώνονται με έναν δίκαιο τρόπο, με θεμητό τρόπο. Εάν μια, ένα αποδεκτικό στοιχείο, για παράδειγμα, προέρχεται από βασανισμούς θα πρέπει να ακυρώνεται και είναι στοιχείο το οποίο συντείνει υπέρ της αθότητας του κατηγορουμένου. Η Επίτροπος κυρία Γιούροβα, σας ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την κυρία Ναταλή Γκρισπέκ και τους συνεισηγητές για την επίτευξη ταχείας συμφωνίας σχετικά με αυτή την οδηγία. Το κείμενο αυτό δεν είναι μόνο ε, μία διακήρυξη αρχών και στόχων έτσι ώστε να καταστεί αποτελεσματικό το τεκμήριο της αθωότητας σε όλα τα κράτη-μέλη. Αντιθέτως θα ενισχύσει το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη και θα προστατεύσει τα δικαιώματα των υπόπτων και κατηγορουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα τεράστιες ανισότητες ως προς την εφαρμογή του τεκμηρίου αθωότητας υπάρχουν στην Ευρώπη και αυτό το αυτό φαίνεται από τις πρόσφατες καταδίκες των κρατών μελών από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το συμβιβαστικό κείμενο που θα ψηφίσετε αύριο είναι καλά ισορροπημένο, βασίζεται στην Ευρωπαϊκή ε, Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιωμάτα και στη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η οδηγία απαγορεύει τη δημόσια αναφορά στην ενοχή, περιλαμβάνει σαφείς κανόνες για το βάρος της απόδειξης, το βάρος της απόδειξης το φέρει η εισαγγελική αρχή και σκόπος είναι να ωφεληθεί ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος. Το δικαίωμα του σιωπάν, το δικαίωμα του να μην ε, ε, ε, εμπλέκει κανείς τον εαυτό του σε με τα λόγια του σε ποινικό κολάσιμα δικείμενα, όλα αυτά προστατεύονται, καθώς και το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να κάνει δύο δηλώσεις. Πρώτον, μια διευκρινήση για το πώς ερμηνεύουμε το κείμενο σε σχέση με το δικαίωμα του Σιωπάν και το δικαίωμα του να μην πει κανείς κάτι που θα το φέρει σε χειρότερη νομικά θέση. Και δεύτερο, το θέμα του βάρους της απόδειξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λυπάται για τη διαγραφή της αρχικής παραγράφου. Ανησυχία μας ήταν η εξής. Από τη στιγμή που υπάρχει το δεκμήριο της αθότητας ήδη στα κράτη-μέλη, είναι σημαντικό στο κείμενο της οδηγίας να γίνεται αναφορά έτσι ώστε όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες για τους εναγόμενους να υπάρχουν. Μιλούμε για αυτό ακριβώς. Ωστόσο, το συμβαστικό κείμενο είναι πολύ ικανοποιητικό. Πιστεύουμε ότι τα πρότυπα αυτής της οδηγίας θα ενισχύσουν το ευρωπαϊκό δίκαιο και θα εφαρμοστούν ως τέτοια. Αυτά καθεφτά αμέσως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυ στην ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών και θα μεριμνήσει έτσι ώστε να εφαρμόζεται σωστά στην πράξη. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκάλ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγήτρια Ναταλή Γκρισμπέκ για την εξαιρετική της εργασία σε ένα πολύ πολύπλοκο και σημαντικό ζήτημα. Το τεκμήριο Θότος αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, θεμελιώδες αρχή στα δικονομικά δικαιώματα και οδηγεί σε δίκαιη δίκη. Επομένως το κείμενο το οποίο θα ψηφίσουμε συμβάλλει πάρα πολύ στο να, έχουμε μια ένα καθεστώς δίκαιη δίκη για όλους τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα απαραίτητα δικαιώματα υπεράσπισης. Είμαστε ικανοποιημένοι από το σερωπημένο αυτό κείμενο. Είναι πολύ σημαντικό να προασπίσουμε τα δικαιώματα τόσο των ύποπτων όσο και των κατηγορουμένων και να ενισχύσουμε τα βασικά δικονομικά δικαιώματα του τεκμηρίου αθεότητας χωρίς να θέτουμε ένα κινδύνο βέβαια την ένωμη τάξη. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε καταλήξει σε σωστά ισορροπημένου συμβιβασμού και μπορούμε να δημιουργήσουμε ελάχιστα πρότυπα για τα δικονομικά δικαιώματα, τα οποία αυτή τη στιγμή αρχίσουν να ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη, θα συμβάλλουν αναμφίβολα στην αποτελεσματικότητα του δικαστικού μα συστήματο παντού στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε κυρία Σίπελ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Μία οδηγία για το τεκμήριο αθεότητας. Γιατί δεν πρόκειται και μια αυτονόητη αρχή του κράτους δικαίου που είναι δρεωμένη στα δικαιακά συστήματα των χωρών μελών. Ναι, παρόλα αυτά από το, από το 2007 έως το 2012 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ε, έκανε 26, πρέπει σε 26 παραβια, διαπίστωση 26 παραβιάσεις σε 11 χώρες μέλη. Ωστόσο δεν είναι αυτή η αρχή η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί. Στι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο ακούσαμε ότι υπήρξαν προσπάθειες να αποδυναμωθεί το δικαίωμα σιωπής και το δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης και έγινε επίσης μια προσπάθεια εκ μέρους του Συμβουλίου να αντιστραφεί το βάρος της αποδείξεως. Αλλά χάρη στην, στις προσπάθειες της συγκεκριάς μας μπορέσαμε να τον εμποδίσουμε και μπορέσαμε να εμποδίσουμε ε, κατηγορούμενοι να παρουσιάζονται ως καταδικαστέντες, με το να μεταφέρονται στην ε, αίθουσα του δικαστηρίου μέσα σε ένα κλουβί ή να φορούν χειροπέδες. Η αναγκαία συνεργασία μεταξύ ε, αστυνομίας και δικαστικών ε, αρχών προϋποθέτει την τήρηση βασικών δικαιωμάτων ε, ναι, ασφαλώς και χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία για το δεκμήριο αθεότητας και για άλλα οικονομικά δικαιώματα και το κείμενο το οποίο έχουμε μπροστά μας συνιστά έναν καλό συνδυασμό. Ωστόσο και η καλύτερη νομοθεσία είναι άχρηστη εφόσον δεν εφαρμόζεται. Και γι' αυτό, στο σημείο αυτό, ναι μεν δεν παρήστε το Συμβούλιο, αλλά πραγματικά αναμένω από τις κυβερνήσεις αυτές, αυτοί και, οι άλλοι και οι λοιποί νόμοι να εφαρμοστούν αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιαντόφσκι. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκρισπέκ για όλη αυτή τη δουλειά που έκανε ε, για την ενίσχυση του τεκμηρίου αθωότητας. Θα έχει θετικό αντίκτυπο η έκθεση αυτή, η οποία ακολούθησε τις αρχές της ε, χρηστής σύνταξης του ορθολογισμού και θα ενισχυθούν τα στοιχεία κλειδιά που είναι τα τεκμήρια αθωότητα στην ποινική διαδικασία των κρατών μελών. Η Πολωνία μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος όταν ελευθερώθηκε η χώρα οικοδόμησε το ποινικό της δίκαιο με βάση το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν θα επανέλθω στα ευεργετικά στοιχεία της έκθεσης που έχουν ήδη αναφέρει οι προλαλήσαντες. Θα πω ότι είμαστε υπέρ της έκθεσης έτσι όπως προέκυψε από τον τριμερή διάλογο. Απορρίπτουμε όλες τις τροπολογίες που παρουσιάζουν κινδύνους, κινδύνους να παραλύσει η ποινική διαδικασία. Και γι' αυτό το λόγο οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές θα στηρίξουν την έκθεση στην μορφή που προτείνει η συγκήτρια, η κυρία Γκρίσπεκ. Δηλαδή, στην εκδοχή που προέκυψε από τον τριμερή διάλογο. Οι τροπολογίες, όπως σας είπα, περιλαμβάνουν διάφορα στοιχεία μη ορθολογικά που δεν εγγυώνται καθόλου την αποτελεσματικότητα της ποινική διαδικασίας. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη η συνέχεια σε αυτή την ιστορία και ελπίζουμε να υπάρξει πρόοδος στο ποινικό δίκαιο και να προχωρήσει και η οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ελπίζω οι εργασίες ε, και για αυτό το κείμενο να προχωρήσουν γρήγορα και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άλμπρεχτ παρακαλώ από τους Πράσινους. Ο κύριος Πάτεν. Αυτή η έκθεση υιοθετεί κάποιες από τις αρχές που υπάρχουν στο αγγλικό common law εδώ και αιώνες. Για παράδειγμα το τεκμήριο της αθωότητας, το βάρος της απόδειξης, το δικαίωμα του σιωπάν, της μη αυτοενοχοποίησης, το δικαίωμα του να παρίσταται κανεί στη δική του δίκη και το καθεξή. Είναι ηρωνικό το ότι το Βρετανικό Κοινοβούλιο έχει εγκαταλείψει αυτέ τι αρχέ γιατί οθέτησε τα ενωσιακά νομικά εργαλεία. Π.χ. το τεκμήριο τη αθωότητας το οποίο βρίσκεται στο αγγλικό δίκαιο για 8 αιώνε. Με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης μπορούμε να παραδώσουμε ένα πολίτη για να μπει φυλακή σε μια ξένη χώρα χωρί να παρουσιαστούν αποδεκτικά στοιχεία σε βάρο του ενώπιον αγγλικού δικαστηρίου. Αυτό ή έρχεται σε ευρύ αντίθεση με το τεκμήριο της αθωότητας. Πρώτο καθήκον των ε, Βρετανών βουλευτών είναι να προστατεύσουν τις ελευθερίες του λαού τους και αντί αυτού μας έχουν προδώσει και ντροπή τους για αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λεμπρετών θα ήταν ο επόμενος, αλλά έχετε μπλε κάρτα, τη δέχεστε. Είστε έτοιμος να απαντήσετε την μπλε κάρτα. Κύριε Μπάτεν, τι δέχεστε? Καλώς. Τότε ο κύριος Ποσπίσαλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα τα όσα είπε ο προλαλής σας. Μα ακριβώ επειδή έχουμε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψη, μπορούμε αυτή τη στιγμή να εκδώσουμε πολίτες προς άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό το ότι έχουμε κάποια ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά την ποινική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να εκδίδουμε πολίτες σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουμε κατά αυτόν τον τρόπο κάποια ελάχιστα πρότυπα. Ναι, αλλά ξέρετε ότι κατά αυτόν τον τρόπο αθώοι Βρετανοί πολίτες έχουν φυλακιστεί σε χώρες όπως η Ελλάδα, ενώ οι άνθρωποι αυτοί ήταν αθώοι. Ενώ αν είχαμε μια σωστή διαδικασία έκδοση, θα είχαμε δει τα αποδεκτικά στοιχεία, θα βλέπαμε ότι δεν υπήρχαν αποδεκτικά στοιχεία και δεν θα είχαν σταλεί οι άνθρωποι αυτοί σε άλλε χώρε. Υπήρχε μια Ευρωπαϊκή Σύμβαση Έκδοση στο παρελθόν, η οποία θα μπορούσε να έχει ισχύσει αντί για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Στην περίπτωση όμω αυτή πραγματικά θα μπορούσε ένα πραγματικό δικαστήριο να εξετάσει πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία και μόνο τότε οι άνθρωποι αυτοί θα αποτελούσαν αντικείμενο έκδοση. Ποτέ πριν και ποτέ σε καμία άλλη περίπτωση. Ο κύριο Λεμπρετόν έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το τεκμήριο θώτας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Η Γαλλία όμως δεν χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσει αυτό το δικαίωμα. Ξέρετε ότι ε, ήδη οι φυστάμενε συνθήκες που είχαμε πριν από τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης πληρούσαν τις απαιτήσει αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε περίπτωση δεν είναι σε θέση να προασπίσει το δικαίωμα αυτό χωρίς να το υπονομεύσει. Το βλέπουμε αυτό και στα πλαίσια της οδηγίας. Το άρθρο 5 λέει ότι μπορεί να αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης και το βάρος αυτό να βαρύνει τελικά τον ένοχο, τον ύποπτο και όχι τις διοκτικές αρχές. Κάτι ακόμα πιο ανησυχητικό το εκτιμώντας 17 χρησιμοποιεί μέτρα καταστολής προκειμένου να έχουμε κάποια αποδεικτικά στοιχεία ή μαρτυρίες από τον ίδιο τον ένοχο, από τον ίδιο τον ύποπτο κατηγορούμενο. Για ποιο λόγο να μην χρησιμοποιήσουμε και τα βασανιστήρια θα έλεγα εγώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση τραπεζών και λομπιστών, δεν καταλαβαίνει τίποτα από ελευθερία. Απέχει πάρα πολύ από τις αρχές της ελευθερίας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Μουσολίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο προλαλής σας είπε ότι στη Γαλλία έχουμε ήδη το τεκμήριο αθότητας, μα και στην Ιταλία υπάρχουν εθνικές νομοθεσίες υπέρ του τεκμηρίου αθότητας, αλλά δυστυχώς παραβιάζεται συνεχώς αυτό το δικαίωμα. Γι' αυτό τον λόγο είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η οδηγία. Και θα ήθελα να πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ισορροπημένα δικαιώματα μεταξύ διοκτικών εισαγγελικών αρχών και υπεράσπισης. Ξέρετε ότι πολύ συχνά εγώ ασχολούμαι στην Ιταλία με περιπτώσεις γυναικών που έχουν αποτελέσει αντικείμενο, έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και πολύ φοβάμαι, πολύ συχνά βλέπω ότι στην Ιταλία οι γυναίκες αυτές έχουν λιγότερα δικαιώματα από τον ίδιο το βιαστή τους τελικά. Θα ήθελα λοιπόν η οδηγία αυτή να αποτελέσει ελάχιστο πρότυπο σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωση πρότυπα τα οποία θα καταφέρουμε στη συνέχεια να βελτιώσουμε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου τελικά να καταφέρουμε να πούμε κάτι το οποίο λέγεται ήδη στην οδηγία. Να έχουμε δηλαδή ένα σύστημα εμπιστοσύνη, ένα δικαστικό σύστημα εμπιστοσύνη παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την εκδίκαση των ποινικών αδικημάτων. και ιδίω όσον αφορά τη διαρροή κάποιων πληροφοριών προς τον τύπο. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αντιμετωπίσουμε. Και όσον αφορά το εντούμπιο προωρέο, το ότι ισχύει η αρχή το εναφιβολία υπέρ του κατηγορουμένου, αυτό είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ισχύει αυτή η αρχή. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ φορέ οι ύποπτοι, οι οποίοι θεωρούνται κατηγορούμενοι κατά τη διάρκεια τη ποινική διαδικασία, προτού καταλήξουμε δηλαδή σε τελεσίδικη απόφαση. κυρία Κινίτση έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Ρισπέκ για την εξαιρετική τη εργασία. Το τεκμήριο θότο αποτελεί βασική αρχή του κράτου δικαίου. Αλλά χωρί να έχουμε ένα κοινό πλαίσιο εγγύσεων, τότε θα παραβιάζεται συνεχώ αυτή η αρχή. Πολύ συχνά βλέπουμε ότι ε, η αμοιβαία αναγνώριση κάποιων τέτοιων θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν προστατεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθεί λοιπόν η οδηγία αυτή να καλύψει αυτέ τι αδυναμίε. Εμεί στην Επιτροπή Λίμπη είχαμε υποστηρίξει την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το τελικό αυτό κείμενο διατηρεί τελικά πάρα πολλά από τα θετικά σημεία τα οποία προσπάθησα και εγώ με τη δική μου γνωμοδότηση να προασπίσω. Ορισμένα ευαίσθητα σημεία, όπω για παράδειγμα το βάρο τη απόδειξη ή η ε, χρησιμοποίηση κάποιων αποδεικτικών στοιχείων, με την ε, χρησιμοποίηση καταστολής είναι ζητήματα τα οποία θίγονται στην οδηγία αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε σε όλα τα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε κοινά πρότυπα. Κατά αυτόν τον τρόπο τα εθνικά συστήματα θα αναγκαστούν να συμμορφωθούν με τα ευρωπαϊκά πλέον πρότυπα. Ο κύριος Τσεκόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, είναι συμβολικό το ότι σήμερα καθόμαστε εδώ και διαπραγματευόμαστε για αυτή την οδηγία, ενώ εσείς η ίδια ξέρετε πολλά. Έχετε προσωπική πείρα για το τεκμήριο της αθωότητας στην τσεχική δημοκρατία. Ο τύπος σας δυσφήμισε και σας κατηγόρησε για δικήματα που δεν διαπράξατε εσείς ποτέ και θέλω να εκφράσω το θαυμασμό μου στο πρόσωπό σας και στην ε, δεοντολογία σας και στη συμπεριφορά που έχετε επιδείξει μέχρι σήμερα. Πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάθε κατηγορούμενο, κάθε, κάθε κατηγορούμενο ως αθώο μέχρι ότου αποδειχθεί η ενοχή του. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνεται αυτόματα. Καμία χώρα δεν θα πρέπει να πράττει διαφορετικά. Πρόκειται για θεμελιώδη κανόνα κάθε ε, ε, ποινικού δικαίου σε οποιαδήποτε ένομη τάξη. Το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη είναι αδιαπραγμάτευτο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει μόνο να στηρίζει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά θα πρέπει να εγγυάται και να επιβλέπει τη συμμόρφωση των ε, κρατών μελών. Ο κύριος Μπούντα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ανησυχώ πάρα πολύ με το γεγονός ότι ε, δεν σεβόμαστε σε πάρα πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ένα από τα δικαιώματα αυτά είναι εκ το τεκμήριο αθωότητος. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να προασπίζεται το δικαίωμα αυτό και να έχουμε και τους απαραίτητους μηχανισμούς για να χορηγούμε αυτό το δικαίωμα σε όλη την ποινική διαδικασία. Ως προς αυτό είδαμε ότι υπολείπονται τα δικαστικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζουν τεράστιες αποκλίσεις. Οι δικαστικές αποφάσεις θα πρέπει να ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να θεωρούνται λοιπόν ισότιμες, να είναι άμεσα αναγνωρίσιμες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να έχουμε μια έντονη δικαστική συνεργασία και στον τομέα αυτό, στην προάσπιση δηλαδή του τεκμηρίου αθότητα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά τη δίκαιη δίκη, κατά τη διάρκεια όλη τη ποινική διαδικασία. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό οποιοδήποτε ύποπτο ή κατηγορούμενο για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα να έχει πρόσβαση σε δικηγόρο κατά τη διάρκεια όλη διαδικασία και το δικαίωμα να επικοινωνεί με τρίτου καθώ επίση και με τι προξενικέ αρχέ τη χώρα του κατά τη διάρκεια τη περίοδου σύλληψη. Το να εγκρίνουμε την οδηγία αυτή ουσιαστικά σημαίνει ότι δίνουμε περισσότερα χέγγια για μια δίκαιη δίκη. Κατά αυτόν τον τρόπο κανεί δεν θα θεωρείται ένοχος προτού ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία. Ο κύριος Ράντεβ έχει το λόγο. Το τεκμήριο της αθότητας είναι μια θεμελιώδης αρχή της δικονομικής ε, διαδικασίας. Εμείς ε, στην Ευρώπη έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να δείξουμε στον υπόλοιπο κόσμο πώς ε, το ποινικό δίκαιο και τα οικονομικά δικαιώματα του κατηγορούμενου θα πρέπει να κατοχυρώνονται. Και πραγματικά ε, θα, είναι να... θα πρέπει το τεκμήριο αθεότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις ε, χώρες μέχρι την τελική εξακρίβωση του κατά πόσο ο κατηγορούμενος έχει διαπράξει το αξιόπινο αδίκημα. Ε, ένα άλλο θετικό στοιχείο της οδηγίας είναι ότι οι δημόσιες αρχές δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουν ένοχο των ε, κατηγορούμενων εκ των προτέρων. Μόνο το δικαστήριο μπορεί βάσει του, των αποδεικτικών στοιχείων να αποφανθεί για την ενοχή του κατηγορουμένου. Ο κατηγορούμενος δεν θα πρέπει να εμφανίζεται ως ένοχος στην ε, κοινή ε, γνώμη. Και ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να περιορίζεται το δικαίωμα ελεύθερη διακίνηση του κατηγορουμένου εφόσον αυτό δεν είναι αναγκαίο τα ελάχιστα δικονομικά δικαιώματα θα εγγυηθούν μια δίκαιη δίκη και την ε, εφαρμογή αμοιβαίου σεβασμού των δικαστικών αποφάσεων της κάθε χώρας. Τώρα έχουμε διαδικασία του Catch Ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος ε, Κέλλη. Προφανώς ε, το τεκμήριο της αθεότητας είναι ένας βασικός πυλώνας της ε, δημοκρατίας ε, και είναι καλό που σέρφουν την προσοχή μας σε αυτό το θέμα ε, σήμερα. Ορισμένες φορές, ωστόσο, είναι δύσκολο να τηρηθεί αυτή η βασική αρχή. Λόγω της οικονομικής ύφασης, ορισμένοι τραπεζίτες, για παράδειγμα, ή και πολιτικοί, ε, δεν είναι καθόλου δημοφιλής και τελικά κατηγορούνται από τα ΜΜΕ ε, και θεωρούνται ένοχοι πριν από την διεξαγωγή της δίκης και πολύ συχνά οι ίδιοι όπως και οι οικοι τους ε, υφίστανται δυσμενείς πεπτώσεις. Ε, πολύ περισσότερο από ότι αν είχαν ε, κρατηθεί σε φυλακές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ενισχυθούν τα δικαιώματα αυτά ε, όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Ο κύριος Χρυσόγωνος έχει το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενίσχυση του τεκμηρίου της αθωότητας του κατηγορουμένου στην ποινική δίκη, την οποία συζητούμε σήμερα, αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση της περαιτέρω κατοχήρωσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. ιδιαίτερα σημαντικό είναι να καταστεί σαφές ότι το τεκμήριο αθωότητας σύμφωνα με την οδηγία αυτή καταλαμβάνει και τις τυχόν παράπλευρες διοικητικές συνέπειες της άσκησης ποινική δίωξης όπως παραδείγματος χάριν την αυτοδίκαιη θέση υπαλλήλου σε κατάσταση αργίας. πρέπει να γίνει δεκτό ότι παρόμοιες ρυθμίσεις των εθνικών νομοθεσιών είναι θεμιτές μόνο όταν πρόκειται για αναγκαία μέτρα εν ώψη του είδους και της φύσης του ποινικού αδικήματος και κάτω από την προϋπόθεση ότι έχουν προσωρινό χαρακτήρα και οι συνέπειές τους έρονται πλήρως σε περίπτωση απαλλαγής του κατηγορουμένου στην ποινική δίκη. η εξαίρεση των διοικητικών διαδικασιών από το τεκμήριο αθωότητας που προβλέπεται στην έκτη αιτιολογική σκέψη οδηγίας αφορά μόνο τις αυτοτελείς ενέργειες των διοικητικών αρχών. Ο κύριος Ποσπισίλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα σημείο μόνο θέλω να θίξω. Νομίζω ότι η εναρμόνιση είναι θετική σε ορισμένες περιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την νομική βάση, αλλά εδώ πέρα τα πράγματα λίγο διαφέρουν και το ξέρει πολύ καλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ ήμουν υπουργός δικαιοσύνη στη χώρα μου στο παρελθόν, ιδίω όταν μεταφέραμε την οδηγία για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα και τότε είχαμε πει ότι όντω θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα έκδοση πολιτών σε άλλη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι κοινοί κανόνε προστασία των πολιτών αυτών. Αυτό σημαίνει κοινά ευθυγραμμισμένα δικονομικά δικαιώματα. Γι' αυτό το λόγο υποστηρίζω την οδηγία αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Αν τελικά οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι να αποτελέσουν αντικείμενο έκδοση σε άλλα κράτα-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα πρέπει να υπάρχουν και κοινά δικονομικά δικαιώματα. Ευχαριστούμε, Επίτροπο Γιούροβα έχει το λόγο. Αξιότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία για το τεκμήριο αθωότητας αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς το να έχουμε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνη ασφάλειας όπως ακριβώς έγινε και με άλλες οδηγίες όπως αυτή του 2010 ή την οδηγία για την ενημέρωση του 2011 ή όπως και η οδηγία πρόσβαση σε δικηγόρο που εγκρίθηκε το 2013. Θα ήθελα λοιπόν να σε ενθαρρύνω όλους να υπερψηφίσετε την έκθεση αυτή αύριο και προσβλέπω στην ψηφοφορία που θα γίνει για την οδηγία, για, τις για τα δικά τα δικονομικά εχέγγυα για τα παιδιά. Έκθεση την οποία εγκρίνετε εσείς πριν τα Χριστούγεννα και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε με τον ίδιο επικοδομητικό τρόπο να διαπραγματευτούμε και μια οδηγία για την νομική αρρωγή. Η κυρία Γκρισμπέκτορ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για να συνοψίσω με δύο λόγια, θα ήθελα μετά τις παρεμβάσεις ε, των συναδέλφων να υπογραμμίσω ότι παρά το ότι ε, υπάρχει εθνική νομοθεσία για το τεκμήριο αθωότητας παρόλα αυτά σημειώνονται καταστρατηγήσεις ε, σε αυτό το δικαίωμα στην Ευρώπη και τα παραδείγματα είναι πολύ άριθμα και έτσι διαβρώνεται αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα. Είναι όμως ένα θεμελιώδες δικαίωμα και απαραίτητο για να αποφύγουμε το αυθαίρετο στη διαδικασία. Είναι ένας από τους πυλώνες της δημοκρατίας. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία, σε αυτή τη στέρεα συμφωνία, μια εποχή κατά την οποία η δημοκρατία και το κράτος δικαίου υφίστανται τεράστιες επιθέσεις ακόμα και εντός ευρωπαϊκού χώρου. Ξέρετε, εγώ είμαι νομικός και με μεγάλη περηφάνεια συμμετείχα σε αυτή τη ε, διατύπωση, σε αυτό το κείμενο. Ε, ο κύριος Λεμπρετόν είπε ότι η οδηγία είναι ατελείωτη και ασαφής, όμως είναι 15 τα άρθρα της οδηγίας μόνο. Ε, νομίζω ότι είναι σύντομη και αξίζει την προσοχή όσων είναι νομική όπως οι υποφαινόμενοι. Συμφωνώ με τους περισσότερους συναδέλφους η οδηγία αυτή έρχεται σε συνέχεια του οδικού χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικονομικά δικαιώματα με σκοπό την οικοδόμηση μιας Ευρώπης την οποία φιλοδοξούμε πολύ. Δηλαδή μια Ευρώπη που θα σέβεται το δικαίωμα της υπεράσπισης το δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του, μια Ευρώπη που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω ε, εκ βάθους καρδίας να ευχαριστήσω τους σκιώδης εισηγητές για την κοπιώδη εργασία τους για την ε, σωστή διατύπωση αυτού του κειμένου. Θέλω να ευχαριστήσω και την Επίτροπο, κυρία Γιούροβα, η οποία από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας πρόσεξε ιδιαίτερα και μας βοήθησε ε, αρκετά. Θέλω να ευχαριστήσω τη Λετωνική Προεδρία και τη Λουξεμβούργια Προεδρία διότι συνεργάστηκαν μαζί μας για την οριστικοποίηση αυτού του κειμένου καθώς και όλες τις ομάδες που δούλεψαν τόσο σκληρά για να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ελπίζω ότι αύριο θα τύχει στήριξη με ευρεία πλειοψηφία η έκθεση αυτή και θα ενταχθεί ε, στον νομικό πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. για τα δικονομικά ε, δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Πέρα τη συζήτηση. Τώρα θα έχουμε κοινή συζήτηση για την εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς. Διαδικαστικό κύριε Μαριά. Ε, αρκετά αργά. Παρακολουθούμε τη συζήτηση εδώ και αρκετές ώρες, προσπαθώντας να συμμετάσχουμε στο ΚΑΤΣΔΙ θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα κάνετε στην επόμενη συζήτηση θα δώσετε μόνο σε τρεις συναδέλφους ή θα κρατήσετε τη διαδικασία catch είναι σημαντικό να το ξέρουμε ούτως ώστε να μην αναμένουμε άδικα. αν να δώσετε μόνο σε δύο τρεις συναδέλφους προφανώς δεν μπορούμε να παραμείνουμε απλά μόνο ακροατές. πέστε μας τι θα κάνετε για να το ξέρουμε. ευχαριστώ. Ναι, ο πρόεδρος αποφασίζει πόσο Catch the Eye θα κάνει, σε πόσους θα δώσει το λόγο και γι' αυτό συνεχίζουμε. Πρόκειται για την έκθεση Ford ε, ε, για τα μέσα ατομικής προστασίας, για την έκθεση ε, για τις συσκευές αερίου και την έκθεση Αντώνιο Λόπεθ Ιστουριτς White για τις εγκαταστάσεις με, σειρ, σειρματόσχημα.